συνεδρίαση. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Άντερσον για διαδικαστικό. You have the floor. Έχετε το λόγο. Αντερσον, you have the floor. Κύριε Άντερσον, έχετε το λόγο.